απόγευμα και λοιπόν το διευθυντικό εγκρίνεται. Τέλος, τρίτη ανακοίνωση. Σύμφωνα με τον κανόνα 105.6, ο πρόεδρος της διάσκεψης των προέδρων με ενημέρωσε ότι δεν εκφράστηκαν ενστάσεις για τη σύσταση της Επιτροπής ΕΚΟΝ να μην εκφράσει ένσταση σε πράξη καταξουσιοδότηση. Εάν εντός 24 ωρών δεν εκφραστούν ενστάσεις από πολιτική ομάδα ή από σύνολο τουλάχιστον 40 μελών, η σύσταση θα θεωρηθεί εγκεκριμένη. Ιδάλλως η σύσταση θα ψηφιστεί και διατίθεται στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας στη σύσταση αυτή. Σας ευχαριστώ και έτσι ολοκληρώνονται οι ανακοινώσεις. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, κάπως καθυστερημένο, είναι μια κοινή συζήτηση για τον προπολογισμό